Alors bonjour, euh, bienvenue à tous et θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω μερικά, μερικές πρακτικές λεπτομέρειες. Ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διερμηνία σε διάφορες γλώσσες, με τις οποίες απαριθμεί η Πρόεδρος, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Καλημέρα σας από την ελληνική καμπίνα, μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε ελληνικά. Έχουμε πολλές γλώσσες, λέει η Πρόεδρος. Μπράβο μας. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι και εγώ μπορώ να μιλήσω στα ισπανικά, πράγμα που θα κάνω άμεσα. Καλή σα ημέρα, καλή, καλώς ορίσατε ε, και εσείς ε, μέλη του πάνελ, ε, αυτοί έγκριτοι ομιλητές που θα μας μιλήσουν σήμερα, αλλά καλώς ορίσατε και εσείς συμμετέχοντες θα ήθελα να πω ότι έχουμε ε, ένα πολύ ε, διαδραστικό πάνελ, ένα πάνελ ε, συνεργατικό και που αποτελείται από ανθρώπους υψηλωτά του επίπεδου και μεγάλης εμπειρίας, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια διάσκεψη σαν τη δική μας, σαν τη σημερινή. και βεβαίως αυτό που με διαβεβαίωσαν ε, οι ομιλητές του πάνελ είναι ότι ε, θέλουν να περιμένουν και ερωτήσεις από εσά. Έχετε την ε, δυνατότητα μέσω εντύπου να ζητήσετε να παρέμβετε και μπορείτε να σημειώσετε το όνομά σας, να το δώσετε στη γραμματεία το έντυπο αυτό. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να ε, προσδοκούμε ότι η συνεδρίασή μας θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αυτό που προσπαθούμε να αναλύσουμε σε αυτήν την διάσκεψη ε, που αποτελεί μεγάλη, ένα μεγάλο εγχείρημα έξυπνο, ευφιές και έγκαιρο και βεβαίως και εξ του Κοινοβουλίου και εξ ονόματος ε, της Ισπανικής Αντιπροσωπείας και όλες της γραμματείες ε, Πραγματικά χαιρόμαστε που είμαστε εδώ ε, και που μπορούμε να δείξουμε ότι η παρατήρηση εκλογών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και παίρνουμε πολύ σοβαρά ακριβώς τη δημοκρατία και παίρνουμε πολύ σοβαρά το ασκήν την πολιτική και επομένως ε, η προώθηση, η ενδυνάμωση της δημοκρατίας ή των δημοκρατιών, ε, ακόμα και οι ανατροπές οι δημοκρατικές ε, στον κόσμο, το κράτος δικαίου, ο, ο, σεβασμός του νόμου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων όντων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δράσεις προτεραιότητας και επομένως αυτή η δράση της συμμετοχής σε παρατήρηση εκλογών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εξού ε, και ε, ο προβληματισμός μας όσον αφορά αυτήν την ιδιαίτερα περίπλοκη δράση. προτεραιότητά μας αποτελεί η δημοκρατία, διότι ε, ακριβώς η πρώτη στην προτεραιότητά μας ε, είναι οι πολίτες ε, και οι συμμετέχοντες στην πολιτεία και ακριβώς θέλουμε να ακολουθήσουμε και να βοηθήσουμε, να είμαστε αρρωγοί στις εκλογικές διαδικασίες αυτών των πολιτών. Γνωρίζομαι ότι υπάρχουν ε, κάποιες αναταραχές οι οποίες είναι αποδεκτές ε, στα πλαίσια μιας δημοκρατίας, αλλά μερικές ε, φορές δεν είναι και απολύτως φυσιολογικές καταστάσεις σε εμπεδομένες δημοκρατίες. Ωστόσο, παρατηρούμε και καταστάσεις περίεργες και σε χώρες οι οποίες αναζητούν ακόμα την οδό της δημοκρατίας, αλλά και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου. Σε ορισμένες ε, χώρες ε, είναι ε, γεγονός ότι η διαφορά ε, από ποια πλευρά βρίσκεσαι, αν είσαι στην πλευρά ε, που κατέχει την εξουσία ή την πλευρά που αναζητά την εξουσία, είναι ο διαχωρισμός πολλές φορές οριακά ακόμα και ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Και σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις χώρες είναι ασταμάτητος, άοκνος αγώνας αυτός της προσπάθειας να επιτύχει κανείς την εξουσία συνεργασία με δημοκρατικά μέσα. Ε, υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ε, σε περιβάλλον ύψης της αντίθεσης ή βίας και εκεί βλέπουμε τι σημαίνει βία, τι σημαίνει μεγάλο επίπεδο βίας, πίεση, κοινωνική βία, πολλές πράξεις ε, ε, εκφοβισμού από πλευράς ε, των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών έτσι ώστε να λύσουν εσωτερικά αλλά και εξωτερικά προβλήματα, τρομοκρατία επίσης, ένοπλες ομάδες κόμματα τα οποία δεν αποδέχονται την έκβαση των εκλογών και το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν άνθρωποι και κόμματα τα οποία είτε δεν δέχονται τα αποτελέσματα, είτε ανατρέπουν τα αποτελέσματα ε, κλπ. Όλες αυτές είναι διαδικασίες μέσα από τις οποίες πρέπει να μάθουμε ε, περισσότερα στοιχεία. Εγώ ως βουλευτής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως έχουσα υπάρξει επικεφαλής διαφόρων αποστολών πιστεύω ότι μόνο μέσα από τη βαθιά γνώση μπορούμε να προωθήσουμε την εργασία την οποία πρέπει να κάνουμε και την εργασία βεβαίως την οποία πρέπει να κάνουν αυτοί τους για τους οποίους ασκούμε την ε, παρατήρηση των εκλογών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού υπάρχουν ε, πολλές ε, οργανώσεις και πολλά μεμονωμένα άτομα τα οποία γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα Διάλογο. όσον αφορά σειράξεις, ένοπλες σειράξεις κλπ. Και Άλλωστε, ο στόχος της σημερινής συζήτησης, της συνεδρίας αυτού του πρωινού, είναι όλοι όσοι έχουν γνώση, όλοι όσοι ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό, να δημιουργήσουν συνέργειες. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τις χώρες και το ύψιστη απόδειξη του σεβασμού είναι η παρατήρηση εκλογών ε, εντός ενός περιπλόκου συστήματος και βέβαια Καλό είναι να διαβάζουμε τα εγχειρίδια πολιτικής και να διαβάζουμε και τις ειδήσει και να διαβάζουμε και βιβλία ή περιοδικά. Αλλά πάντα η πραγματικότητα ξεπερνάει αυτά που ε, υπάρχουν μέσα στα βιβλία. Γι' αυτό λοιπόν μέσω της εγκύτητος ε, ε, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση και όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν καθημερινά στο πετσί τους αυτή την κατάσταση, αυτή τη βία, πρέπει και εμείς με απτό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κατάσταση. Εγώ ήμουνα στην IT ε, ε, σε επικεφαλής ομάδας παρατήρησης εκλογών και να σας πω ότι δεν υπάρχουν την ημέρα των εκλογών δημόσια μέσα μεταφοράς. Ε, πολύ Και αυτό γίνεται ε, διότι, δεν, διότι συχνά ε, υφίστανται βανδαλισμούς την ημέρα των εκλογών τα μέσα, τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε μια χώρα τόσο φτωχή όσο η IT δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι οι ψηφοφόροι ένα μέσο για να πάνε να ψηφίσουν και ε, ε, πρέπει να περπατήσουν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Ωστόσο στην Αιτή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό ανθρώπων με αναπηρία στη χώρα αυτή ε, ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών και συστήματος υγείας περίπου ανύπαρκτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορεί να κινητοποιηθεί η κοινωνία ε, στην IT ε, ε, τη στιγμή που θα πρέπει για να πάει κανείς στα εκλογικά κέντρα να περπατήσει ώρες και ώρες. σε μια χώρα μάλιστα που οι φυσικές συνθήκες, οι κλιματικές είναι τρομερές. Έξι το πρωί χτυπάει ήδη ο ήλιος πολύ δυνατά στην Αϊτή. Και σας επαναλαμβάνω, επειδή επιτέθηκαν πάρα πολύ συχνά και έκαναν βίες πράξεις και βανδαλισμούς στα μέσα μεταφοράς, την ημέρα των εκλογών δεν υπάρχουν μέσα. Ε, αυτά τα απλά πράγματα, αλλά και τα πολύ πιο σοβαρά, πρέπει εμείς να ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Και για αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Η βία σε πολλά μέρη του κόσμου είναι δυστυχώς σχεδόν διαρθρωτική και Επομένως και, η, πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να ειδωθεί εκτός αυτού του πεδίου των βία, το, ε, της βίας. Ε, ενώ υπάρχουν σε άλλες, ε, και άλλες περιπτώσεις όπου η βία ε, είναι συγκυριακή και αφορά μονάχα την εκλογική διαδικασία. είναι σημαντική η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Ε, όπως και το θέμα των βιωτοτήτων είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, είτε είναι διορθωτικό είτε ε, συγκυριακό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την κατάσταση, να αναλάβουμε ευθύνη κατά κάποιο τρόπο της κατάστασης. Ωστόσο, εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε ανεξάρτητοι αλλά βεβαίως μπορούμε να ε, ε, ε, συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου, οι οποίοι ασκούν τη διαμεσολάβηση και γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. όσον αφορά τις διαδικασίες της παρατήρησης εκλογών. Ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης εμείς αποκτούμε όλο και περισσότερα εργαλεία. Ωστόσο, πρέπει κάθε φορά να έχουμε υψηλό πολιτικό ε, φρόνημα κατά κάποιο τρόπο, υψηλό ε, πολιτικό περιεχόμενο ε, στην δουλειά μας. Οι τεχνικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα, θα τολμούσα να πω ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο. Ahora necesitamos que los políticos lo hagan casi tan bien como los técnicos. <laughs> Ε, έχουμε εδώ μερικού ε, τεχνικούς, ε, πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε ακριβώς αυτές τις τεχνικές ομάδες από τις οποίες και εμεί, οι βουλευτές, άνδρε και γυναίκες μαθαίνουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν θέλω να πάρω χρόνο από τους έγκριτους καλεσμένους μας και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μοχαμέτ Τσάμπας, ο οποίος είναι ειδικό ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων ε, για την ε, Δυτική Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ. Πρόκειται για άνθρωπο μεγάλης εμπειρίας σε περιοχές ε, σειράξεων. Ε, πριν ε, ήταν ειδικό απεσταλμένος για την ειρήνευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Αφρικανική Ένωση στο Νταρφούρ. Έχει ασχοληθεί πολύ με τη Λιβερία καθώς επίσης και με την ακτή του Εντεβαντοστού. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρυτάτη εμπειρία του, θα ήθελα να ρωτήσω, κατά την άποψή σας, ποια είναι τα σημαντικά σημεία, τα σημεία κλειδιά σε μια ε, εκλογική διαδικασία που μπορούν να οδηγήσουν σε βία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, στα πλαίσια της προληπτικής διπλωματίας, της έγκαιρης διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης, ούτως ώστε ε, σε όλο τον εκλογικό κύκλο να μπορέσουμε με συγκεκριμένο τρόπο να συμβάλλουμε στην ειρήνη ή στην επίλυση ε, των ε, σειράξεων και όχι να ρίξουμε λάδες στη φωτιά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε ε, επαφή με τις αρχές και με τους υποψηφίους. Αυτά θα θέλαμε να μας πείτε και σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ εγώ. Η θητεία της υπηρεσίας μου, του γραφείου των, του ΟΗΕ για τη Δυτική Αφρική και το Σαχέλ, βασίζεται στην εργασία που γίνεται στην ε, πρόληψη, κυρίως στην ε, πρόληψη βίαιων ε, συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά βεβαίως και για την πρόληψη βίων συγκρούσεων στην, χώρα, στην επικράτεια της ευθύνη μας. Και βεβαίως υπάρχουν και θέματα διαμεσολάβησης με τα οποία ασχολούμαστε και η δημιουργία ειρηνικού περιβάλλοντος στη, στα κράτη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κινητοποιεί, τι θα μπορούσε να κινητοποιήσει την βία σε, μια, σε ένα εκλογικό περιβάλλον. Χτες στις συζητήσεις ένα μέλος του Κοινοβουλίου της Κένιας έθεσε ένα θέμα και ρώτησε αν το θέμα είναι μόνο οι εκλογές ή αν πρέπει τελικά να διορθώσουμε την πολιτική. Το ίδιο θέμα το ε, ανέφερε και ο Πατ Μέρλο που είπε για την ε, Κένια και παραθέτω αυτό που δεν πήγε καλά στην ε, Κένια δεν ήταν ότι απέτυχε η τεχνολογία, είναι ότι απέτυχε η πολιτική. Ένα κομμάτι λοιπόν, ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το σωστό πολιτικό περιβάλλον, τους σωστούς πολιτικούς θεσμούς και να υπάρχει βεβαίως και μια ε, ήρεμη εκλογική διαδικασία. Αν, ας πούμε, οι θεσμοί στην χώρα δεν μπορούν να οργανώσουν αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες, τότε πρέπει να περιμένετε ότι οι χαμένοι προφανώς θα ε, αντισταθούν και δεν θα αποδεχτούν το αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών από τα θεσμικά όργανα. Δεν θα πω εγώ περισσότερο γι' αυτό, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι εδώ στο πάνελ που θα μιλήσουν ε, με λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Ένα ε, ήρεμο περιβάλλον σημαίνει ότι θα πρέπει και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να μπορούμε να προλάβουμε τα hot spots, τα προβληματικά σημεία που μπορεί να υπάρξουν πριν φτάσει κανείς καν στην περίοδο της εκλογικής διαδικασίας. Στην Κάνα, ας πούμε, συνεργαζόμαστε στενά για να ενισχύσουμε το Εθνικό Ειρηνευτικό Συμβούλιο να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις. Γιατί αν δεν γίνει αυτό σε επαρκές επίπεδο, οι εκλογές που ούτως ή άλλως είναι πολύ έντονες και πολύ ανταγωνιστικές περίοδοι, πολύ φορτισμένες πολιτικά, μπορούν όντως να καταλήξουν σε βίαιες συγκρούσεις. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σε χώρες ώστε να υπάρξει εθνική ομόνια, εθνική συνένεση. Ας πούμε στη Δυτική Αφρική, στο Τόγκο και στην Κάμπια γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Μόνο αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν ε, ε, όριο στις θητείες. Το Τόγκο ε, προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα και υπάρχουν βεβαίως και πολλές διαδηλώσεις που, που γίνονται στους δρόμους για το θέμα αυτό. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πάμε σε εκλογές χωρίς να λυθεί το πρόβλημα αυτό θα δημιουργήσει όντως πολλές πιθανότητες βίας. Και γι' αυτό η υπηρεσία μου συνεργάζεται και με άλλους εταίρους, δίνει την στήριξη που χρειάζεται στον διάλογο που γίνεται στο Τόγκο, έτσι ώστε να υπάρξουν και οι συνταγματολόγοι που μπορούν να υποστηρίξουν τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που ελπίζουμε ότι πριν το τέλος του τρέχοντος θα γίνουν, ώστε να υπάρξουν θητείες συγκεκριμένες για τις κυβερνήσεις στο Τόγκο να μπορούν ε, να ε, λαμβάνουν μέρος και γυναίκες. Όλα αυτά τα θέματα, εάν λυθούν, θα μειώσουν τις πιθανότητες εντάσεων και συγκρούσεων στο Τόγκο. Και στην Κάμπια το ίδιο. Από την ε, ανάληψη της κυβέρνησης από τη νέα κυβέρνηση, Ουσιαστικά υποστηρίζουμε μια πρωτοβουλία που ε, ονομάζεται «Διατηρούμε την ειρήνη». Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και σε συνταγματικά θέματα, να σχεδιάσουν δηλαδή το νέο σύνταγμα για τη νέα Γκάμπια. Ένα από τα θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές είναι η επανεισαγωγή των ε, ορίων θητείας. Αυτά είναι λοιπόν τα σημεία που θεωρούμε ότι μπορεί να κινητοποιήσουν τη βία και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις χώρες που τα αντιμετωπίζουν. Επίσης, η πρόληψη της βίας και η διατήρηση της ειρήνης. Πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές, όχι μόνο εκλογικές επιτροπές όπως είπα, αλλά και το δικαστικό σύστημα Πολλές φορές ε, χρειάζεται κατάρτιση στοχευμένη, συγκεκριμένη για να δημιουργηθεί ε, ακριβώς ε, περισσότερη γνώση σε όλο, στο δικαστικό σώμα από τα κατώτερα δικαστήρια μέχρι τον Άριο Πάγο έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να διαχειρίζονται, να διεκπεραιώνουν υποθέσεις που σχετίζονται με διαφορές εκλογικού χαρακτήρα. Γιατί όταν δεν λύνονται τα θέματα αυτά, πάλι υπάρχει πιθανότητα κατά τη διάρκεια της εκλογική εκστρατεία να δημιουργηθούν ε, συγκρούσεις. Κάτι άλλο που θέλω επίσης να πω είναι ότι η υπηρεσία μου συνεργάζεται με κράτη-μέλη για να δημιουργήσει μια αρχιτεκτονική εθνικής ειρήνης. Ούτε ο ΙΕ, ούτε η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ούτε οι τοπικές ε, ε, ε, οργανώσει μπορούν να είναι πάντα σε όλες τις χώρες και σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια αρχιτεκτονική εθνική ειρήνη σε κάθε χώρα και βεβαίω θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρμόζεται στις εθνικές, στα εθνικά χαρακτηριστικά. Στην Κάνα υπάρχει αυτό και σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ καλά οργανωμένο και σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η Νιγηρία πρόσφατα δημιούργησε μια εθνική επιτροπή εκλογών. Πέρασε τη σχετική πράξη και ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά που θα γίνουν εκλογέ θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Χρειάζεται λοιπόν μια εθνική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ε, ακαδημαϊκοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αναγνωρίσιμοι Νιγηριανοί και αυτό θα γίνει και σε επίπεδο περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική τους λοιπόν η θητεία θα έχει να κάνει με την καταγραφή προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις και αντιδράσεις. Και βεβαίω θα πρέπει από μόνοι του να κάνουν την προσπάθειά του σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό για να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Αν υπάρχουν αυτού του είδου οι αρχιτεκτονικέ, αυτού του είδου οι δομέ, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και το ε, σωστό ε, περιβάλλον κατά τη διάρκεια των εκλογικών ε, διαδικασιών. Και εφόσον θα υπάρχει και αποδοτική λειτουργία της διαχείρισης των εκλογών και υπάρχει επαγγελματισμός και διαθεσιμότητα και από τις υπηρεσίες ασφάλειας, θα υπάρξει μείωση της βίας κατά τη διάρκεια της, των εκλογών. Και η υπηρεσία μας ε, συνεργάζεται στενά με όλους αυτούς τους εταίρου, γιατί οι εταιρικέ σχέσεις για μα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εταιρικέ σχέσεις με τις περιφερειακές ε, οργανώσεις, με την ΕΚΟΑΣ, και με, την, ε, με τις οργανώσεις της Λιβερίας, της Σιέρα Λεόνε. Χτες κάναμε κάποιες διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο για, για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, την κυρία Σαμάτη, για να οργανώσουμε μια κοινή αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΚΟΑΣ και του ΟΗΕ στην Ιγυρία, γιατί πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση. Θα πάμε λοιπόν εκεί ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εμπλακούν σε αυτή την συζήτηση. Και βεβαίω και όλοι οι υποψήφοι των βασικών δύο πολιτικών κομμάτων. Πρέπει και αυτοί από την αρχή της διαδικασίας να μπουν στο παιχνίδι για να ε, δεσμευθούν ότι θα εξάγουν ε, εκλογικές διαδικασίες, εκλογικές εκστρατείες ε, ήρεμες, χωρίς προβλήματα, χωρίς βία. Και θα συνεργαστούμε φυσικά ώστε να υπάρξει και ένα εθνικό φόρουμ όπου θα υπογραφεί ένας κώδικας δοντολογίας για τις εκλογές στην Ιγερία γιατί όπως ξέρετε οι εκλογές στην Ιγυρία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Ιγυρία. Έχουν να κάνουν, αν πάνε καλά, σημαίνει καλά αποτελέσματα και για τη Δυτική Αφρική, αλλά και συνολικά για την Αφρική. Αν πάνε άσχημα όμως και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο μπορεί αυτό να έχει στη Δυτική ε, Αφρική, αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Ε, σταματώ εδώ.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 En fin, es otra persona con muchísima experiencia eh, no solo teórica, sino Πρόκειται για ένα άτομο με ε, μεγάλη εμπειρία, γνώστη ε, του πεδίου δράσης. Ε, όπως σας είπα προηγουμένως είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη ε, που ακριβώς έχει στόχο την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών με στόχο την ειρήνη. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτό ε, το συντονιστικό εργαλείο βάσει της εμπειρίας σας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια, πρακτι... κάποια παραδείγματα βελτίστων πρακτικών ε, από πλευράς της πράξης των ΕΕ και των ε, ομάδων. Επίσης, πρόληψη συγκρούσεων στα πλαίσια των νέων πολιτικών ηγετών που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Τι μπορεί να γίνει πόση σημασία μπορεί να έχουν τα τμήματα νεότητας των πολιτικών κομμάτων σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, πιστεύετε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ε, την συνεργασία, το συντονισμό με άλλες κοινέ αποστολές, με άλλους διεθνείς φορείς. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η ικανότητά μας μέσω αυτού του τρόπου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Ε, να μοιραστώ μαζί, μου την, μαζί σας την τεχνογνωσία που βέβαια είναι ε, και πολύ διευρυμένη σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν αρχικά και για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκλογική παρακολούθηση, ε, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και όταν στρέφονται όλα τα βλέμματα του κόσμου ε, σε μια εκλογική διαδικασία πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο τουλάχιστον αξιοπιστία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Και νομίζω ότι όλες οι αποστολές ε, εκλογικής παρατήρησης ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Εγώ έχω πολιτικό υπόβαθρο, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, ε, γιατί πολύ συχνά οι διπλωμάτες ρωτούν αν οι πολιτικοί έχουν κάποια οποιαδήποτε σημασία και αξία. Εμείς αυτό που ξέρουμε σαν πολιτικοί είναι πώς να κάνουμε εκστρατείε κάποιε φορές και πώς να ιδρύσουμε ένα κόμμα. Εγώ εργάστηκα στο Σουντάν και στον Ταρφούρ και ήταν το πιο σύνηθες ερώτημα. Πώς κάνει κανείς μια εκστρατεία. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Είναι διαφορετικά βέβαια τα πράγματα σε διαφορετικέ εκστρατείε στη Φιλανδία και στον Ταρφούρ, αλλά οι βασικέ αρχέ είναι κοινέ. Είναι πολύτιμη αυτή η γνώση. Και το να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο άλλος για το πώς θα κάνεις την εκστρατεία, πώς θα επικοινωνήσεις με το κοινό σου, πώς θα δημιουργήσεις μια κυβέρνηση συνασπισμού και να μην ακολουθεί την τακτική του ε, ο νικητής τα παίρνει όλα. Αυτό έχει να κάνει και με τα διάφορα τι πολιτικές εμπειρίες που υπάρχουν. Και αυτό έχει να κάνει και με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη, αλλά και ε, για διάφορα ε, πολιτικά ιδρύματα και που αξιοποιούν την ευκαιρία που υπάρχει ε, και γίνεται αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων που υπάρχει σε αυτή την πολιτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω. Πριν περάσουμε στην εκλογική διαδικασία, φυσικά και πρέπει να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική διαδικασία, συμφωνία. Θυμάμαι όταν εργαζόμουν με τον Νότιο Σουδάν, ο... κάποια από τα πολιτικά κόμματα είπαν ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποιες περιοχές, γιατί δεν είναι ασφαλής για εμάς για να κάνουμε και την εκστρατεία μας. Και δυστυχώς οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να διασφαλίσουν ε, ακριβώς ε, την ασφαλειά μας. Μπορεί δηλαδή ήδη να βρισκόμαστε σε προεκλογική φάση, αλλά να μην υπάρχει ασφάλεια. Αυτό πρέπει να έχει γίνει από πριν, στην ειρηνευτική διαδικασία. Συρία, Ιεμένη, Λιβύη, σε τέτοιες χώρες απέχουμε βέβαια πάρα πολύ από το να έχουμε κανονικές εκλογές. Βέβαια μπορούμε συνεχώς να αισιοδοξούμε και να ονειρευόμαστε για το πώ θα γίνουν οι εκλογέ εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα, συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, με τα κλίματα πολέμου. Στη Συρία έχουμε τον Ασάντ, υποψηφίου, ε, υποστηρικτέ του. Ξέρετε τώρα πώ είναι αυτά τα πράγματα, πώ είναι τα διλήμματα. Έχουν να κάνουν με αποτρόπε πράξεις που έχουν λάβει χώρα και συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα. Και εδώ αναφέρομαι και στη Λιβύη και στην Ιεμένη και την περίπτωση της Ερυθρέας παρακολουθώ εκτός συναγκής, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια επισκεφτόμαι συχνά αυτή τη χώρα. Φέτος έγινε ένα θαύμα. Γιατί και άνοιξαν τα σύνορα με την Αιθιοπία, αλλά κάποιοι ήρθαν και μου είπαν, παρεμπιπτόντως είμαι και μέλος του Κοινοβουλίου. Και αυτό δεν το έχω ακούσει εδώ και χρόνια στην Ερυθρέα, να είναι κάποιος βουλευτής. Αλλά τώρα κάτι, κάτι αλλάζει. Βλέπω ότι έχει συμβολική αξία. Ε, είναι ένα όνειρο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και εδώ εκλογές. Και βέβαια, όταν εξομαλυνθούν οι σχέσεις με την γειτονική χώρα στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας και αυτό θα ανοίξει το δρόμο και για τις ε, συνήθεις παραδοσιακές εκλογικές και πολιτικές διαδικασίες. Ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω εδώ είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Σε ό,τι αφορά τι κεντρικές αφρικανικές δημοκρατίες, μπορεί κάποιοι να... μάλλον για την κεντρική αφρικανική δημοκρατία, μπορεί κάποιοι να λένε ότι οι κάτοικοι του Τσάντ θα πρέπει να φύγουν. Κάποιοι λένε πόσο καιρό είναι εδώ η υπήκοοι του Τσάντ, μόνο 100 χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουν αντίστοιχη συζήτηση με την ε, μειονότητα Ροχίνγκια. Πόσο καιρό είναι εδώ, μόνο 100 χρόνια ήρθε η ώρα να φύγουν. Και βέβαια δεν γίνεται να έχουμε ε, κανονικές πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες σε ένα τέτοιο κλίμα όταν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με τις μειονότητες. Πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα πριν γίνουν εκλογές. Αναφέρετε και εσείς, Πρόεδρε, πρέπει να μιλήσουμε και για τις γυναίκες εδώ. Όταν έχουμε να κάνουμε με τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές και πώς πρέπει να τις στηρίξουμε, υπάρχουν πολλές κουλτούρες όπου υπάρχουν διακρίσεις κατά των γυναικών. Ευτυχώς στην Αφρική έχουμε κάποιες θετικές εξαιρέσεις όπου είναι υψηλή η συμμετοχή των γυναικών, ακόμα και ηγούνται σε ορισμένε περιπτώσει του πολιτικού προσκυνείου. Η Λιβερία είναι ένα καλό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλε περιπτώσει όπου οι γυναίκε αποκλείονται από το πολιτικό βίο. Και όταν περνάμε από εμφύλιο πόλεμο, φτάνουμε μετά στις εκλογικές διαδικασίες, ε, πολύ συχνά εκεί οι γυναίκες αποκλείονται. Επομένω, το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το 2035 είναι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα το ψήφισμα 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας μιλά ε, και για τον ρόλο των νέων σε αυτή την πολιτική διαδικασία. Πέρυσι ήμουν στο Αφγανιστάν και ήρθα αντιμέτωπο με μια εξαιρετική κατάσταση. Ε, γνώρισα ανθρώπους που παλιότερα ήταν με τους Ταλιμπάν, όπως ο κύριος Μουταμπακίλ, που σήμερα ζει στην Καμπούλ. Το μήνυμά τους ήταν ότι τώρα χρειάζονται βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Πολύ ενδιαφέρον είπα εγώ, γιατί εσείς δημιουργήσατε τις ταραχές σε αυτή την κοινωνία. Όχι, χρειαζόμαστε βοήθεια κατά του ISIS ε, που στρατολογεί ε, νέους από τα σχολεία και το πανεπιστήμιο στην Καμπούλ και τους στέλνει στη Συρία. Ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή η ένδειξη. Και ξέρετε ότι οι νέοι πιο εύκολα στρατολογούνται και δραστηριοποιούνται και στον ένοπλο αγώνα και πρέπει να τους διδάξουμε τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας και τη σημασία της συμμετοχής σε εκλογικέ διαδικασίες. Και θα μείνω εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, bueno, ahora tenemos... Πολύ ωραία. Προσπαθούσα εδώ να στείλω ένα tweet σχετικά με το συνέδριο, την αίθουσα, listening room κλπ. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί, μπερδεύομαι. Ε, λοιπόν, έχουμε τώρα ε, έναν άνθρωπο εγνωσμένου κύρους, τον κύριο Jason Carter, πρόεδρο του κέντρου Carter, Ως πρόεδρος της Επιτροπής Χορηγών ε, αυτού του κέντρου, έχει συμμετάσχει πολλές φορές ε, σε παρατηρήσει εκλογών και όχι μόνο. πρόκειται για ένα κέντρο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις χώρες ε, στις οποίες δρά. Πιστεύετε ότι η παρατήρηση εκλογών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της βίας και επιπλέον πιστεύετε ότι θα πρέπει αυτή ακριβώς η μείωση της βίας να αποτελεί μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ε, τμήμα της εντολής ε, στην ε, διάρκεια της παρατήρησης εκλογών. Και συνδέω με αυτό το ότι η ανάγκη ε, ανεξαρτησίας ε, είναι οπωσδήποτε ε, εγγενός, ε, αποτελεί συγγνώμη, εγγενός τμήμα της παρατήρησης των εκλογών. Πρέπει κανείς να είναι αμερόληπτος και ανεξάρτητος. Και τέλος... Πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές οι ε, δικές μας δηλώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από την αντιπολίτευση σε ορισμένες περιπτώσεις, λέω, έτσι ώστε να ε, καταφερθούν κατά του αποτελέσματος, να αμφισβητήσουν ε, το αποτέλεσμα των εκλογών. Με ποιο τρόπο πιστεύετε, μάλλον, είναι δυνατόν αυτού του είδους η παρέμβαση να προκαλέσει βία μετά τις εκλογές. Άρα, συνοψίζω, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της ειρήνης πριν την εκλογική διαδικασία και πώς μπορούμε να αποφύγουμε η δικιά μας συμμετοχή να έχει συμβάλει στην αύξηση της βίας μετά τις εκλογές. Uh, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα με τόσο εγκεκριμένου ε, προσκεκλημένους και φυσικά και με ευρύτερη συμμετοχή. Εκτιμώ αυτή την ε, ευκαιρία και τα όσα είπαν και συνάδελφοι και χθε για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Όταν μιλούμε για εκλογικές διαδικασίες και τις ε, δυσκολίες που έχουμε, όχι μόνο με εκλογικά συστήματα, αλλά και με την πολιτική συμπεριφορά που ε, βρίσκουμε σε διάφορες δημοκρατίες, εγώ ομολογώ ότι κατάγομαι από τις ΗΠΑ που ίσως έχει γίνει ε, παράδειγμα προς αποφυγή πλέον από πλευράς πολιτικής συμπεριφοράς. Το κέντρο Κάρτερ έχει συμμετάσχει σε αποστολές σε πάνω από 100 ε, αποστολές παρακολούθησης και σχεδόν πάντα υπήρχε η πιθανότητα ε, διένεξης. Εκεί δηλαδή όπου υπήρχε μεταβατική φάση προς μια δημοκρατία ή όπου η δημοκρατία έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον υπάρχει ε, ενδεχόμενο να ξεσπάσουν βία φαινόμενα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η διεθνή παρατήρηση εκλογών έχει πολύ σημαντικό ρόλο να δραματίσει ό,τι αφορά ε, την αποφυγή της βίας. Για να απαντήσω λοιπόν το πρώτο ερώτημα, μπορώ να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου μπορούμε να συγκεράσουμε την προϋπόθεση οι διεθνείς παρατηρητές να είναι αντικειμενικοί και ουδέτεροι με την ιδέα ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ειρηνευτική διαδικασία. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες ημέρες. Πρώτον, λοιπόν, από τους πιο σημαντικού τρόπους με τον οποίο με, με τις μπορούμε να φέρουμε ή να διατηρήσουμε την ειρήνη είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε αυτό το σύστημα. Είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα πρέπει βέβαια να εδράζεται στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια. Εμείς λοιπόν ως εκλογικοί παρατηρητές είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια και κάποιες φορές μπορεί να είναι και δύσκολη η αλήθεια. Μπορεί και να αποσταθεροποιείς τα πράγματα. Όμως μπορούμε αυτή την ειλικρίνειά μας να τη συνδυάσουμε και με σεβασμό προς τον λαό. Με κατανόηση της δημοκρατίας. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο που μιλούσε προηγουμένως για την αξία των πολιτικών. Και παρότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να αποτελούν και παράδειγμα προσωπική σε κάποιε περιπτώσει, κάποιε άλλε φορέ όμω είμαστε και ένα παράδειγμα προ μίμηση. Όταν οι εκλογικοί παρατηρητέ συνομιλούν με του ηγέτε για το τι νόημα μπορούν να, να πάρουν οι εκλογικέ διαδικασίε είναι ότι το μονοπάτι της ειρήνης είναι το μονοπάτι της πολιτική. Γιατί ποια είναι η εναλλακτική ε, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα είναι να βγούμε από το πολιτικό σύστημα όπου και πάλι ξεφεύγουμε. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει μόνο εμπιστοσύνη στον, στη λειτουργία του εκλογικού συστήματος, αλλά ότι και στο μέλλον εσείς ως μειονότητα ή ως ε, ε ιτημένο πολιτικό κόμμα θα μπορείτε να ξαναβρείτε τις δυνάμεις σας και να συμμετάσχετε στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ένα λοιπόν από τα πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς ως εκπρόσωποι του Κέντρου Κάρτερ και άλλοι που ε, συμμετέχουν στις εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας τους είναι ότι μπορούμε να καθίσουμε με μια ομάδα και να πούμε «Ωραία, χάσατε αυτές τις εκλογές, τι θα κάνετε τώρα, εκστρατεία για τις επόμενες εκλογές». Με αυτή τη μορφή, με αυτή τη συνεργασία με τους νέους, όπως είπε και ο συνάδελφος, από τις πιο καλές συναντήσεις που έχω κάνει στην καριέρα μου ήταν με μια ομάδα νέων στη Λιβερία, που είχαν ενδιαφέρον να μάθουν πώς μπορούν ε, να επανέλθουν. Όμως εντός του πολιτικού συστήματος, όχι εκτός. Θέλει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να δουν πώς μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στον πολιτικό στίβο. Αυτό χρειάζεται συζήτηση με απεσταλμένους και από τα δικά μας ιδρύματα και από τις ΗΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ότι μπορεί δηλαδή να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούν να συνεχίσουν την εκλογική αυτή διαδικασία. Που είπε και ο κύριος Σάμπας προηγουμένως. Οι προεκτάσεις μπορούν να έχουν για τους ιτημένους οι διαδικασίε εντό του πολιτικού προσκυνείου είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν ότι όλο ο κόσμο του παρακολουθεί και ότι έχουν και πολιτική ευθύνη εναντί του κόσμου, αλλά από την άλλη ότι γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο σύστημα. Έχει να κάνει λοιπόν και με τις πολιτικές δομές που έχει να κάνει και με την πολιτική ευθύνη και λογοδοσία, αλλά και την δύναμη, την ενδυνάμωσή τους, ότι δηλαδή θα τους πιστέψουμε αν βγουν και νικητές της εκλογικής αναμέτρησης. Άλλα δύο ζητήματα θα ήθελα να θίξω. Και ίσως εδώ και η χώρα μου είναι σημαντικό παράδειγμα. Εγώ κατάγομαι από την Τζόρτζια ε, και ήμουν, κατέβηκα και σε εκλογέ για τη θέση του κυβερνήτη πριν από τέσσερα χρόνια και έχασα. Έχουμε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων στην Τζόρτζια με πολύ μεγάλη οικονομία, ε, με πολύ μεγάλο αεροδρόμιο. Μπορεί να έχετε περάσει κιόλα πηγαίνοντα προ τι ΗΠΑ. Όμω τώρα έχουμε ε, και ένα ιστορικό υπόβαθρο ε, φιλετικών διακρίσεων, διακρίσεων κατά των γυναικών τον επόμενο μήνα για πρώτη φορά μία γυναίκα από, που προέρχεται από μειονότητα είναι βασική υποψήφια. Είχαμε δικαστική απόφαση που έλεγε ότι ε, τα μηχανήματα που θα ακολουθήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε για τις εκλογές ε, δεν είναι ασφαλή μπορούν να χακαριστούν και ότι μετά τις εκλογές δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστώσουμε κατά πόσο ε, όντως υπήρξε χακάρισμα ή όχι. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε χωρίς να υπάρχει πραγματικός φόβος ε, για βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καλό σύστημα. Ούτε ότι αν πάμε στην Κένια και στην Λιβερία εμείς θα τους πούμε πόσο πρέπει να κάνουν τις εκλογές. Όμως σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι και να χάσει κάποιο όποιος ιτηθεί σε εκλογέ, ε, θα παραμείνει εντός του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής δομής. Θα αλλάξουμε βέβαια αυτά που πρέπει να αλλάξουμε, θα αλλάξουμε τα μηχανήματα, αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα. Το τελευταίο που ήθελα να πω, που είναι κρίσιμη σημασία για μένα, είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. η εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα και στο πολιτικό μέλλον έναντι ενός μέλλοντος που έχει να κάνει με τη σύγκρουση απαιτεί οι μειονότητες να πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συνασπισμούς. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα και σε μια δημοκρατία, οι μειονότητες δεν έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν πολιτική ισχύ. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι αυτή η οικοδόμηση συνασπισμών είναι εξαιρετικά σημαντική σε μέρη όπως η Μιανμάρ, όπου όλα τα βασικά πολιτικά κόμματα έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο συνασπισμού. Εκεί πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναλάβει αυτό το καθήκον και να δώσει έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Γιατί ακόμα και αν, αν υπάρχει ειρήνη, δεν είναι σταθερή, είναι ευάλωτη. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στις εθνικές δομές ειρήνης και ότι ο κόσμος όχι μόνο θα πρέπει να εμπιστεύεται την εκλογική διαδικασία, αλλά και το πολιτικό σύστημα, ε, την πολιτική ως μέσο επίλυσης ε, κρίσεων και συγκρούσεων στο μέλλον και το κέντρο Κάρτερ εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται σε αυτό το πλαίσιο και ο παππούς μου ε, γνωρίζει πραγματικά ε, την αξία του να ητάται κανείς σε μια εκλογική διαδικασία και εγώ συνεχίζω και αυτό το έργο. Όμως εκτιμώ τη δυνατότητα που μου δίνεται να είμαι εδώ σήμερα και περιμένω και τα ερωτήματά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, και μία παρατήρηση εκλογών για τη Γεωργία. Ναι, ναι, φυσικά. Ωραία. Η επόμενη ομιλήτρια είναι μία γυναίκα. Εκπροσωπεί το Διεθνές Κέντρο Angie Brooks. Ονομάζεται Ιβέτ Σεσόμ Μπουρέ. Είναι από την ε, Λιβερία, δηλαδή από την ίδια χώρα που ήταν η Angie Brooks, ε, η μόνη ε, γυναίκα ε, από την Αφρική, η οποία, υπήρξε, η οποία προείδρευσε ε, τη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία ε, ασχολείται με την ενδυνάμωση των γυναικών τόσο στη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών, αλλά και εν γέννη στη διάρκεια των πολιτικών διαργασιών. Και έχει δημιουργήσει ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων ε, που αφορούν τις γυναίκες ε, και που ε, κινητοποιείται σε ενδεχόμενες σειράξεις προ των εκλογικών διεργασιών. Η πρώτη Situation Room δημιουργήθηκε για τις εκλογές του 2011 στη Λιβερία και έκτοτε στην Σενεγάλη, στη Σιέρα Λεόνε, στην Ουγκάντα, στην Ιγερία κλπ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας μιλήσετε για τον αντίκτυπο που έχει η εργασία σας και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην μείωση της βίας, να αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο όχημα προς την μείωση της βίας ε, εν ώψη εκλογικών διεργασιών. Ε, ποια μπορεί να είναι επίσης η συνεργασία ανάμεσα σε μια αποστολή παρατήρηση εκλογών που κάνουμε εμείς και ένα δικό σας crisis room. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, ο, και οι δύο να δουλέψουμε ε, στην ίδια τροχιά, έτσι ώστε να συμμετάσχουν οι γυναίκες, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα ε, με ασφάλεια να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογικές διεργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. for this opportunity, for θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ευκαιρία που μας δίνετε ε, σε εμά τις ε, γυναίκες της Αφρικής ε, να συμμετάσχουμε σε αυτό το έγκριτο πάνελ και να συναντηθούμε με ανθρώπους σημαντικούς και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι εμείς οι Αφρικανές γυναίκες δεν φοβόμαστε πλέον. Έχουμε γίνει ατρόμητες βγαίνουμε από τα σπίτια μας και βγαίνουμε και από την ήπειρό μας και παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Δεν την αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια των πολιτικών, δεν την αφήνουμε στα χέρια των ανδρών, την παίρνουμε τη ζωή μας εμείς στα χέρια μας εμείς οι Αφρικανές γυναίκες. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί. Ε, το Women's Situation Room λαμβάνει όλα αυτά ε, ε, πολύ σοβαρά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα συνεχές υπόβαθρο βίας στην ε, Αφρική πέρα από ταξινομήσεις ε, ε, μπορούμε να φτάσουμε από την απλή βία μέχρι την γενοκτονία περνώντας ενδιάμεσα στάδια την βία στο σπίτι, την βία εντός του ζευγαριού κλπ. Και αυτό που κάνει το Women's Situation Room είναι να αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες της Αφρικής. Όχι τις μορφωμένες, όχι αυτές που έχουν σπουδάσει, ε, αλλά κυρίως το αντίθετο. Αυτές που βρίσκονται πραγματικά στο πιο κάτω σημείο ε, της ε, ταξινόμησης, ας πούμε, και που ε, είναι ε, γυναίκες ε, οι οποίες ζουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συνθήκες άθλιες μέσα σε εγκληματικές ομάδες, σε γκάγκς που κοιμούνται σε νεκροταφεία. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας ενδιαφέρει περισσότερο γιατί πιστεύουμε ότι αν σταθεροποιηθούν αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας θα σταθεροποιηθεί η κοινωνία στο σύνολό της και η χώρα μας και οι χώρες γενικά. Γιατί ξέρετε υπάρχουν ε, και οι, ε, καλοθελητές ε, που δίνουν λίγα χρήματα σε νέα παιδιά ή σε νέες γυναίκες και τους λένε πήγαινε ε, κάνε αυτή την κίνηση για να αποσταθεροποιήσεις την, την κατάσταση και το κάνουν για λίγα χρήματα. Εμείς τους βγάζουμε από τα νεκροταφεία και τους δίνουμε σπίτια για να ζήσουν και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτοί οι νέοι μπορεί από τη μία πλευρά να προκαλέσουν χάος ή από την άλλη πλευρά να προκαλέσουν ε, την ε, ειρήνη ε, και δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να τους προκαλέσουμε χάος και εμείς τους λέμε νομίζετε ότι η μάνα σας σας είχε 9 μήνες στην κοιλιά της για να καταντήσετε έτσι. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί για να, να τον κάνετε εσείς χαοτικό με τις ενέργειές σας. Εμείς στο Situation Room έχουμε ε, ε, κάνει πολλές ε, κινήσεις ε, για την ε, παρατήρηση εκλογών και για την ε, μείωση της βίας ενώπιον των εκλογών. Είμαστε οι πρώτοι που οργανώσαμε πορεία για το θέμα αυτό. Ο κύριος Τσάμπας, και θέλω να τον ευχαριστήσω εδώ, μια και είναι παρόν, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, και μάλιστα στην Κάνα ήρθε στο λεγόμενο gang room, ε, το, την ομάδα των εγκληματικών οργανώσεων, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο gang room, ε, γιατί καταλαβαίνετε εμείς προσπαθούμε να έχουμε έναν οργανισμό, συγγνώμη, έναν μηχανισμό άμεσης ανταπόκρισης. Εμείς σε αυτό το gang room έχουμε μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων, έχουμε τους επικεφαλείς τους, λαμβάνουμε τηλέφωνα τηλέφωνα εκείνη την ώρα και απαντούμε επί τόπου. Ήρθε λοιπόν στο gang room και ε, άρχισε να τους μιλάει. Whole room erupts. Και τους μίλησε στη γλώσσα τους και έμειναν με ανοιχτό το στόμα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πριν ε, θορυβούσαν και, και πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Και τους ρωτήσαμε τι κάνατε μέχρι τώρα για την ειρήνη. Και είπε ένας ε, όταν ε, είπε ένα σήκωσε το χέρι του και είπε «Μα την ώρα που ήρθε ο κύριος Τσάμπα στο δωμάτιο και άρχισε να μας μιλάει, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να βγούμε από τα γκέτο, ότι, υπάρχει, ότι έχουμε δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που ε, μοιραία μας οδηγεί στην βία». Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Χαίρομαι επίσης ότι, που είναι εδώ η Τζιν Λάμπερτ που ηγήθηκε ε, της ε, ε, αντιπροσωπείας σε ένα άλλο σημείο που είχαμε Women's Room. Είσαστε κι εσείς σε αυτό το Women's Room. Την ενημερώσαμε αυτήν και την αντιπροσωπεία της. Και ξαφνικά ακούσαμε από την τηλεόραση ότι ένας από τους ε, υποψηφίους ε, των ε, εκλογών στη Σιέρα Λεόνε ότι ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικού γιατί φοβόντουσαν ότι υπήρχαν άνθρωποι με όπλα γύρω του και ξαφνικά μπήκε στο δωμάτιο, στο crisis room η γυναίκα του και είπε βοηθήστε μας γιατί μιλήστε τους. Και πραγματικά ε, συνεργαστήκαμε τότε και μπορέσαμε να ε, χαμηλώσουμε τους ε, τόνους. Ξέρετε, εάν απλά σηκώσει το τηλέφωνο και προσπαθήσεις να μιλήσεις με όλους τους υπόλοιπους φορείς και τους πεις «Είμαστε εδώ», μιλάμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου, βλέπουμε όπλα ή δεν βλέπουμε όπλα, τότε ε, μπορούμε να βοηθήσουμε ε, και στην προκείμενη περίπτωση ε, ήρθαν οι αστυνομικοί και έψαξαν την περιοχή και εν πάση περιπτώσει ξαφνικά Είδαμε μια περίπτωση ότι προσπαθούσαν οι αστυνομικοί να πιάσουν τον ε, Μαχάμα και του είπανε, κουνάγανε ένα χαρτί μπροστά του και του λέγανε ότι εμείς έχουμε ένταλμα σύλληψης και είπε ο Μαχάμα θέλουμε να το δούμε. Και ε, ε, γύρισε ο Μαχάμα και κοίταξε εμένα και μου είπε Πραγματικά είναι ένταλμα αυτό. Ε, και ξαφνικά αναρωτηθήκαν όλοι, μα ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ε, ε, ελέγχει. Αλλά δεν ήταν τελικά ένταλμα σύλληψης. Και Γύρισε λοιπόν ο Μαχάμα και είπε αποφασίσαμε να μην εκτελέσουμε αυτήν, μάλλον γύρισε ο αστυνομικός και είπε αποφασίσαμε να μην εκτελέσουμε αυτήν την ε, εντολή σύλληψης και φύγανε τελικά ε, γιατί εμείς προστατέψαμε τον υποψήφιο, τον άντρα αυτής της γυναίκας. Everybody leaves because I start chasing them outside the building και ε, ε, ε, βγήκαμε έξω από την αίθουσα και ήταν εκεί συγκεντρωμένε γυναίκες από την Σιέρα Λεόνε και πραγματικά προστατέψαμε τον άνθρωπο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η διαδικασία ειρηνευση περνάει και μέσα από πολύ απλά πράγματα, αλλά περνάει και μέσα από τις γυναίκες. Η έγκαιρη, ε, ε, η έγκαιρη παρέμβαση των γυναικών μπορεί πραγματικά να ε, είναι αποτελεσματική. Έχουμε έχουμε βεβαίως και δυνάμεις ασφαλείας που προσπαθούν έτσι ώστε οι εκλογές να λειτουργήσουν καλά. Υπάρχουν ε, και ε, παρατηρητές και ομάδες παρατήρησης εκλογών, αλλά εγώ θα ήθελα περισσότερη παρέμβαση από πλευράς αυτών των ομάδων, περισσότερη δράση, παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Ε, εάν μια ομάδα ε, έρχεται απλά ε, και καταγράφει πέντε πράγματα ε, ως παρατήρηση εκλογών και μετά σηκώνεται και φεύγει, μία τρύπα στο νερό κάνουμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Και μετά μας αφήνεται. Μας αφήνουν όλοι. Θα πρέπει, θα πρέπει κάποιος να βρίσκεται επί τόπου και να καταπραίνει τους φόβους και να λέει έχεις τον νόμο με το μέρος σου και προχώρα. πρέπει να βοηθήσουμε ε, με την παρουσία μας και να βοηθήσετε με την παρουσία σας τις επιτροπές ε, εκλογών να καταλάβουν ότι πρέπει οι εκλογές να γίνονται με ε, σωστό και αμερόληπτο και διαφανή τρόπο. Free, fair and transparent. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας για τις εκλογές ελεύθερες δίκες και διαφανείς ε, και πρέπει να ξεπεράσουμε και ε, ε, την αντιμετώπιση που έχουμε πολλές φορές και γιατί να μιλήσω εγώ με σένα και γιατί να σε λάβω υπόψη μου. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος της κοινωνίας. Κοιτάξτε, εμάς μας ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε από πολύ χαμηλά. Και όταν μιλάμε για βία στη διάρκεια των εκλογών, το τονίζω, δεν θα πρέπει να δείτε μόνο την κατάσταση από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω. Και εμείς έχουμε ακριβώς αυτό το είδος της εμπειρίας. Εμείς κάνουμε αυτό το είδος της ε, διπλωματίας από τη βάση προς τα πάνω. Και ε, είναι σημαντικό να μπορούμε να σηκώσουμε, να έχουμε τη δύναμη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να ζητήσουμε κάτι ή να αποτρέψουμε κάτι. Και πρέπει βεβαίω να έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Μερικέ φορέ πρέπει απλά να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Και να του πούμε πώ έχει η κατάσταση, γιατί μερικά πράγματα δεν τα ξέρει ενδεχομένω. Μία επίσκεψη στην αγορά, ας πούμε, μπορεί να έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ε, γιατί εάν μια γυναίκα ε, μαζί με κάποιο άλλο έγκριτο μέλος της κοινωνίας ε, της χώρας πάει στην αγορά ή κινηθεί και μιλήσει με άλλες γυναίκες και ξέρουν και οι υπόλοιπες γυναίκες ότι θα λειτουργήσει καλά το σύστημα, ότι τα παιδιά τους δεν θα πεινάσουν, ότι τα κορίτσια τους θα πάνε στο σχολείο, τότε πραγματικά ότι θα έχουν περίθαλψη ε, τότε ε, πραγματικά ε, αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα που μια καθημερινή απλή γυναίκα θέλει να ακούσει. Αυτά την ενδιαφέρουν και δεν θέλουμε αυτά τα θέματα να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγοράς ψήφου. Να σας πω και κάτι άλλο. Ε, οι άνθρωποι που έχουν ε, μηχανάκια στην Αφρική και που ε, κυκλοφορούν πολύ είναι η καλύτερη πηγή πληροφορίας. Ξέρουν ανα πάσα στιγμή τι συμβαίνει στην Ήπεθρο. Ξέρουν ανα πάσα στιγμή τι συμβαίνει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρουν αν ετοιμάζεται να ξεσπάσει βία κάπου. Motorcycles of Africa. Είναι και αυτή μια ομάδα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Bueno, eh, Πρόεδρος, όλες οι παρεμβάσεις ήταν εξαιρετικές. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα. Βλέπω εδώ ότι από την αίθουσα έχουμε ε, πολλούς που ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην μακρηγορήσετε έτσι ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Εγώ θα ήθελα όλοι να μπορέσουν να μιλήσουν, να έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα ερώτηση-απάντηση. Νομίζω ότι είναι καλύτερα και είναι και πιο άμεσο και όχι να μαζέψουμε πολλές ερωτήσεις και μετά μια συνολική απάντηση, αλλά γρήγορα όμως. Η Μαρίζα Ματίας, η συνάδελφός μου, έχει πρώτη το λόγο. Είναι βεβαίως βουλευτής του Κοινοβουλίου από την Πορτογαλία. Ε, ε, και εκείνη έχει υπάρξει σε πολλές ε, περιπτώσεις επικεφαλής παρατήρηση εκλογών, τελευταία στις, στην Ονδούρα. Μαρίσα. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέρονται τόσο ακούσαμε από τους ομιλητές, όμως υπάρχουν ακόμα μερικά ερωτήματα. το μία λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ε, καταστάσεις από την ε, Μέση Ανατολή μέχρι τις Ονδούρες. Δεν είναι ίδιες οι εκλογικές παρατηρήσεις. Δεν μιλάω για το τι γίνεται μετά με τις επιπλοκές που υπάρχουν στο εκλογικό και πολιτικό σύστημα, αλλά ισχύει με αυτό που είπατε για τις εκλογές που ξεκινούν πολύ νωρίς ε, το πρωί και με τις χώρες που δέχονται αυτή την εκλογική διαδικασία ως μια ειρηνευτική διαδικασία. Στις Ονδούρες ε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά γιατί εκεί υπάρχει ε, δομική βία συνεχούς έντασης και όταν δεν έχει ξεκάθαρος ε, πόλεμος ε, και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ειρήνη. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που ανέφερε η Έλενα. Πώς οι εκλογές, οι αποστολές μάλλον παρατήρησης, ιδίω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή συγκρούσεων. Να οδηγήσουν στην ειρηνική διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων. Σε ό,τι αφορά την εντολή αυτών των ε, αποστολών, γιατί και εμεί έχουμε συγκεκριμένη εντολή, δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε, ή πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ουδέτεροι. Επομένω, ε, ενώ θα σεβόμαστε λοιπόν αυτή την εντολή, πώ μπορούμε από την άλλη να σα βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί είπαν και οι προηγούμενοι μιλητέ ότι στις Ονδούρες μείνατε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει, γιατί ήταν πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα και αν είχαμε φύγει υπήρχε κίνδυνος ε, μεγαλύτερης αστάθειας. Όμως, η εντολή μας μας περιορίζει από την άλλη. Και με αυτή την εντολή εμείς δεν μπορούμε να εργαστούμε ε, σε ό,τι αφορά την επίλυση συγκρούσεων. Μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη διαχείριση της σύγκρουσης, αλλά μέχρι εκεί. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ της σταθεροποίησης και της σταθερότητας. Μπορούμε να συμβάλλουμε στη συνέχιση της σταθερότητας, αλλά η σταθεροποίηση δεν αποτελεί τμήμα της δικής μας εντολής. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία πρέπει να εργαστούμε εμείς όταν εξετάζουμε νέα ενδεχόμενα νέων δυνατοτήτων για τις ε, αποστολές εκλογικής παρατήρησης. Δεν στρέφουμε προς κάποιον ε, από τους ομιλητές πιο συγκεκριμένα. Όλοι θα έχουν, φαντάζομαι, κάτι να πούν, κάτι να σχολιάσουν. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε. Ε, Νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει ο κύριος Κάρτερ να ξεκινήσει να απαντάει. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Το κέντρο Κάρτερ δεν υποστηρίζεται από κάποια κυβέρνηση και αυτό είναι το καλό. Ένας τρόπος λοιπόν για να σας απαντήσω είναι να σας πω ότι υπάρχουν εταίροι που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν πολλές φορές να κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, άλλους εμπλεκόμενους και η στήριξη που δίνουν είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε χώρες όπως η Ονδούρα ή το Ανατολικό Τιμόρ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς ε, την ε, ισχύ και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, μια δύναμη που μπορεί να σταματήσει διάφορες ε, διαδικασίες. Και το θέμα αυτό είναι να αξιολογήσει κανείς τη δημοκρατία, την αξιοπιστία που θα έχει στο μέλλον αυτή η δημοκρατία. Το να είναι λοιπόν εκεί παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό στοιχείο αυτής της ανάλυσης. Ακόμα και αν καμιά φορά είναι ενοχλητικό γιατί θέλει κανείς να κάνει περισσότερα από μπορεί όταν είναι επιτόπου. Αλλά αυτή η σημαντική πτυχή των αποστολών είναι ότι όσο πιο πολύ μπορούν να είναι αυτές οι αποστολές σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη η βοήθειά τους. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις όπου το κέντρο Κάρτερ, ας πούμε, είχε ομάδες ε, για μήνες ή για χρόνια σε μια χώρα μέχρι να φτάσει η μέρα των εκλογών και έτσι είχε πολύ περισσότερες ε, δυνατότητες να, ε, να, καταγράψει τα σημεία ας συγκρούσεων όπως έλεγε ο κύριος Τσάμπας πιο πριν. Αλλά βεβαίω πάντα ο παρατηρητή πρέπει να σέβεται την εντολή του. Πρέπει όμω να χρησιμοποιεί και την ε, γνώση που έχει. Όταν μιλά με ένα τέτοιο τρόπο ή όταν μιλά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο μια συγκεκριμένη στιγμή, από τη δική του την οπτική, πρέπει να ξέρει ότι θα συμβεί το εξή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πολιτικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εντάσεις, να χρησιμοποιήσουμε την επικοινωνία που έχουμε ως πλατφόρμα αποστολής εκλογικής παρατήρησης για να βρούμε ουσιαστικούς τρόπους να αλλάξουμε τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό, όπως είπατε και εσείς, αλλάζει δραματικά από χώρα σε χώρα. Ο κύριος Χάβης το έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εξαιρετική ερώτηση. Εγώ θα απαντήσω για την Ονδούρα, γιατί α, παρακολουθώ την σχετική υπόθεση Μπέρτα Κάσερες. Α, ήμουνα μάλιστα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και υπόθηκε ότι το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, υπάρχει κάτι εγκρυπτό, Υπάρχουν ε, μυστικές ε, οργανώσεις ε, που παρεμβαίνουν. Αυτό ήταν πραγματικά πολύ ανησυχητικό και ήταν σημαντικό όταν το συζητήσαμε και στην, με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία και τον πρέσβη εκεί. Είχαμε έναν πρέσβη ο οποίος ήταν ανοιχτό για όλες τις μειονότητες και είδαμε τι ρόλο μπορεί να παίξει η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκλογική παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα πορίσματα που είχε συλλέξει κατά τη διάρκεια της ύπαρξης εκεί, της αποστολής και στην Ονδούρα. Εγώ ήθελα να πάω στις περιοχές των συγκεκριμένων μειονοτήτων. Μου είπανε μην πάτε, είναι επικίνδυνα. Ούτε η αστυνομία δεν πάει εκεί, δεν τολμάει. Εγώ πήγα και οι άνθρωποι εκεί μου είπαν να επιτέλους κάποιος ήρθε. Περιμένουμε να έρθει ένας άνθρωπος εδώ και 10 χρόνια. Όταν λοιπόν ε, μπορεί κανείς να φανταστεί μια ε, μειονότητα που είναι άγρια και ζει στο, στην ύπεθρο κρυμμένη από όλου και πάει και τη δει τελικά βλέπει ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια αυτά. Πρέπει ακριβώς να πάμε στα μέρη που δεν μας επιτρέπουν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σας ε, κατευθύνω προς άλλη κατεύθυνση με την απάντησή μου. Ο κύριος Τσάμπας έχει το λόγο. Um, να πω ότι θεωρούμε ότι οι εκλογές είναι μια συνεχής διαδικασία από την προεκλογική ε, εκστρατεία μέχρι την ημέρα των εκλογών και μετά τις εκλογές. Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωνόμαστε ε, σε όλη την περίοδο και όχι μόνο στην περίοδο των εκλογών. Και βεβαίω μετά τις εκλογές όταν κανείς προσπαθεί να δημιουργήσει ειρήνη, σταθερότητα στη χώρα. Εμείς δεν κάνουμε παρατηρήσει όσο ε, πρέπει να πω. Το δικό μας το ενδιαφέρον είναι να δούμε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση, της Αφρικανική Ένωσης, άλλων οργανώσεων και θα μα ενημερώσουν αυτές οι ε, εκθέσεις για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε με τους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς, με τις εκλογικές επιτροπές, για να υπάρχει μια συνέχεια στην ενίσχυση της χώρας βεβαίως. Όταν μια χώρα έχει περάσει από ε, συγκρούσεις, από κρίσεις, προφανώς θα έχει δυσκολίες. Ακόμα και χώρες που δεν έχουν περάσει από τέτοιες κρίσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις εκλογές. Οπότε παίρνουμε την έκθεση και μπορούμε να δούμε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τι λέει η έκθεση και να δούμε πώς από κοινού μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ χαίρομαι με το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στη Δυτική Αφρική. Αυτό λέω στις διάφορες χώρες που επισκέπτομαι. Ότι παρατηρώ ότι σε κάθε επόμενη εκλογή τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι στην προηγούμενη. σε προηγούμενε εκλογέ ε, πέθαναν α πούμε χίλιοι άνθρωποι. Το 2015 για παράδειγμα στην Ιγυρία. Μπορεί να πέθανε και χίλιοι άνθρωποι μάλιστα μετά τις εκλογές, επειδή οι εκλογές ε, έγιναν με σχετική ηρεμία. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και επίση ε, υπάρχει η ισότητα όπλων όλο και περισσότερο τελικά. Από τις τελευταίες 12 εκλογικές αναμετρήσεις, η 9, τις 9 τις κέρδισε η αντιπολίτευση. Συνέβη, μπορεί να μην το παρατηρήσαμε, αλλά συνέβη, που σημαίνει ότι όντως ε, υπάρχει ισότητα δυνάμεων. Τα κόμματα γίνονται πιο επαγγελματικά, γίνονται πιο αποδετικά, πιο αποτελεσματικά. Και βεβαίω όλα αυτά προκύπτουν και από τι ε, εκθέσει που έχετε υποβάλει εσεί μετά, τι αποστολέ παρατήρηση ε, εκλογών. Προφανώ δεν περιμένουμε οι βρουβουλευτέ ε, να έρθουν να μείνουν τρει εβδομάδε. Η δουλειά σα δεν σα επιτρέπει να τόσο, τόσο πολύ χρόνο, αλλά είναι σημαντικό που έρχεστε. Εγώ σα ενθαρρύνω να συνεχίσετε να το κάνετε. Bueno, decidía cómo repartía el ε, Ενώ προσπαθούσα να δω πώς θα μοιράσω το χρόνο, ε, ε, μου έφτασαν άλλες 10 αιτήσει ε, για λήψη για χρονομιλίας ε, και τι να σας πω, θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω. Έχουμε περίπου 30 λεπτά ακόμα, 30 λεπτά για αυτή τη συνεδρία. Έχουμε περίπου 20 εγγεγραμμένους μιλητές, το λέω, έτσι ώστε ε, να προσπαθήσετε να πείτε ό,τι θέλετε μέσα σε ένα, ένα μισή λεπτό, έτσι ώστε να μπορέσουν και τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν. Ε, γιατί εάν ε, υποβληθούν όλα τα ερωτήματα και μετά στις 11 σας πω τώρα τελείωσε πρέπει να φύγουμε, δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν τα μέλη του πάνελ. Συνοπτικά λοιπόν και συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθώντας. Για ένα λεπτό ή ακόμα και λιγότερο, ο κύριος με πιέρα Τζονί Κουαμέν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από το, την κοινωνία των πολιτών ε, και το παρατηρητήριο βελτίστων πρακτικών ε, από την ακτή του Ελεφαντοστού. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την εμπειρία που έχουμε εμείς. Ε, ξέρετε ότι από το 2002 και μετά το 2011 είχαμε κρίσεις στην χώρα μου. Το 2002 αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να οργανώσουμε την κοινωνία των πολιτών ε, σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες ε, πήγαμε και ε, οργανώσαμε, εγκαταστήσαμε επιτροπές επιβα επαγρύπνησης και ειρήνης κυρίως στην κοινότητα ΣΕΝΤΕΑΟ γιατί ξέρετε ότι έχουμε υποδεχθεί ε, αυτήν την ομάδα εμείς. Δουλέψαμε λοιπόν ε, όλοι μαζί έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε όλοι να αποδεχτούμε ο ένας τον άλλον. Τα καταφέραμε και σε δέκα περιφέρειες της ακτής του Ελεφαντοστού έχουμε εγκαταστήσει επιτροπές οι οποίες λειτουργούν μέχρι τώρα και δημιουργήσαμε και τον κώδικα δεοντολογίας των υποψηφίων πολιτικών και με τον τότε Γενικό Γραμματέα Μπανκιμούν ε, συνεργαστήκαμε ε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό το παρατηρητήριο κοινωνίας των πολιτών, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω. Έχουμε δουλέψει καλά, έχουμε προχωρήσει πολύ όσον αφορά ε, την διαβούλευση, όσον αφορά τις εκλογικέ διαδικασίες με, τις, με τους μεγάλες πολιτικούς σχηματισμούς. Δουλεύουμε επίσης ε, με τη Διακομματική Επιτροπή ε, και έχουμε ε, εγκαταστήσει πάνω από 80 επιτηρητές σε ολόκληρη την χώρα που έχουν και την δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα να καταρτίζουν τις νεολαίες των κομμάτων. Και ε, μαζί λοιπόν πηγαίνουμε επί τόπου και μιλάμε στα μέλη των κομμάτων. Να σας πω ότι... Α, πρέπει να σταματήσετε. Ναι, ε, έχουμε τώρα τοπικές εκλογές ε, με εσωτερική βία γιατί προετοιμάζεται με τον τρόπο αυτό η εκλογική διαδικασία του 2020 και εμείς δουλεύουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να σταματήσει η βία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μακ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ τον Μηχανισμό Εξωτερική Πολιτική, που έχει σημαντικό ρόλο να γνωρίσει ό,τι αφορά την οργάνωση των αποστολών εκλογική παρατήρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, θέλω να σταθώ περισσότερο στην πρόληψη των συγκρούσεων και τι κάνουμε με αυτόν τον μηχανισμό σε ό,τι αφορά την συμβολή μα στην σταθερότητα και την ειρήνη. Κάνουμε μια συζήτηση σήμερα για το πόσο θα πρέπει να παραμένουν οι αποστολές ε, στο μέρος της αποστολής. Είναι σημαντικό οι αποστολές αυτές να ακολουθούν λίγο τον παλμό ε, της εκλογικής διαδικασίας. Γιατί κάποιες ε, φορές ε, μπορούν και οι εκλογικέ αξίε να χάνουν, οι αποστολέ να χάνουν την ε, αξία του. Να περιμένουν λοιπόν ε, οι αποστολέ, αλλά να βασίζονται και σε άλλου φορεί και παράγοντε. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν ορισμένα πρακτικά παραδείγματα και εμείς τα στηρίζουμε σε άλλες πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα στο Μαλί προσφάτως. Είναι απλά αυτά τα πράγματα, αλλά ήθελα να τα επισημάνω. Είναι σημαντικό με τα δικά μας προγράμματα να ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους φορείς, εάν μπορούμε, πριν από τις εκλογές. Και εδώ, με αυτό δεν εννοώ τα επιμέρους πολιτικά κόμματα, ούτε μόνο τις πολιτικές ελίτ, αλλά και τους μοτοσυκλετιστές που αναφέρατε προηγουμένως. Να σταθώ και αυτό πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε και πριν και μετά από την εκλογική αναμέτρηση. Πολλές από τις ε, πρωτοβουλίες που υποστηρίζουμε, για παράδειγμα στη Ζιμπάμπουε, αλλά και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, συγγνώμη, στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι σημαντικό να παραμείνουν ε, και εκ των υστέρων. Επίσης σημαντικό είναι να στεκόμαστε και στις εθνικές πρωτοβουλίες και στην οικειοποίησή του σε εθνικό επίπεδο. Όμως θα πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Να μην ακολουθούμε και το κυρίαρχο πολιτικό μήνυμα στην κάθε χώρα, γιατί έτσι μπορούμε να χάσουμε ε, τις μειονότητες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, παράδειγμα, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν θα ψηφίσουν ή τουλάχιστον όχι σε επαρκή επίπεδα, εάν δεν αμφισβητήσουμε τις κυρίαρχες ιδέες. Κάτι τελευταίο τώρα, για την ασφάλεια. Λαμβάνει όλα ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις αυτό το ζήτημα και πολύ συχνά πλέον μα ζητούν να, παρέμβουμε. Στη Λιβύη, για παράδειγμα, αυτό έχει να κάνει την πραγματική σωματική ακαιρεότητα του, ε, του εκλογικού συμβουλίου. Πολύ συχνά όμως πλέον έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα κυβερνοασφάλεια. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, το βλέπουμε τώρα αυτό. Ευχαριστώ. Την ώρα, Σοράγια Πόστ. Η Σοράγια Πόστ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, σοσιαλίστρια, ε, μέλος της Επιτροπής ε, Κοινωνικών ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Και στην ομιλήτρια που εκπροσωπεί τις ε, γυναίκες της Αφρικής. Πραγματικά βλέπω τη δύναμη που πηγάζει από μέσα σας και νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο αυτό θα δούμε και βλέπουμε ότι μας λείπει η δύναμη των γυναικών. και σε ό,τι φορά το πρακτικό σκέλος, όχι μόνο το θεωρητικό. Εγώ είχα πάει στην ε, αποστολή στην Κένια. Ήθελαν οι γυναίκες να ξεκινήσουν ένα σχέδιο δράσης στο Κοινοβούλιο. Δεν έλαβε την ε, πλειοψηφία, αλλά ήταν ένα πολύ ισχυρό και πολύ καλό σχέδιο δράσης. Συζητούσα λοιπόν μαζί τους ε, τα ζητήματα της πολιτικής εκπροσώπησης και μου ανέφεραν δύο ζητήματα. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, πολύ μεγάλη έλλειψη εδώ, για τις ε, υποψήφιες εκλογές. Και το θέμα της ασφάλειας. Όταν πηγαίνουν για να κάνουν την εκλογική του εκστρατεία ή ακόμα και όταν πηγαίνουν να ψηφίσουν, δεν είναι ασφαλής. Επομένω, ίσω ο κύριο Χαβίστε μπορεί να απαντήσει. Πώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για αυτά τα ζητήματα. Φυσικά, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την περίοδο και πριν από τι εκλογέ αλλά και μετά τις εκλογές. Και το επόμενο ερώτημα. Δεν βλέπω ε, και πολλές γυναίκες διαμεσολαβήτριες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Το 1325 λοιπόν, εντάξει, υπάρχει, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Ήμουν και στην Κολεμβία ε, για το δημοψήφισμα σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική διαδικασία και συνάντησα ΜΚΟ, γυναίκες και μου είπαν ότι ήταν από τις πρώτες ε, φεμινιστικές ενευτικές διαδικασίες ε, στην, ε, στον κόσμο. Γι' αυτό και ήταν και επιτυχής. Αλλά ακούγοντας τους Κολομβιανούς σήμερα, υπάρχει φόβος. Και υπάρχει και έλλειψη δράσης της διεθνούς κοινότητας τι προσπαθούμε να κάνουμε τελικά, γιατί όλες αυτές οι αγροτικές περιοχές που έτσι κι ποτέ δεν είχαν αναπτυχθεί. Έτσι έχει κατάσταση σήμερα στην Κολομβία. Και κάτι ακόμα. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ε, κοιτάξτε, αν ο καθένας κάνει τέσσερα ερωτήματα, υποβάλλει τέσσερα ερωτήματα, τι να σα πω τώρα, δεν μπορώ. Ε, ε, James Hamsar από την ε, ομάδα εκλογικής παρατήρησης του Μαλάουι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Όλα όσα μας είπατε είναι πολύ ωφέλιμα για εμάς. Ένα ερώτημα. Μιλήσατε για το 50 συν 1. και ότι υπάρχει δυστυχώς ο κίνδυνος ε, της βίας. Ποια είναι όμως τα ωφέλη πραγματικά του 50 συν 1. Υπάρχουν, υπάρχουν και αρνητικές προεκτάσεις. Ξέρω ότι υπάρχει το οικονομικό σκέλος, για παράδειγμα. Σε μια χώρα όπου εξαρτώμεθα από διάφορους εταίρους ε, για οικονομικούς λόγους. Ποιες είναι οι προεκτάσεις για την καταμέτρηση. Μία από τις ε, τροποποιήσεις ε, του, μάλλον μία από τις τροπολογίες ενός νομοθετήματος ήταν ε, ε, το 50 συν 1, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε. Ξέρουμε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο και πρέπει να το υλοποιήσουμε. Ε, προετοιμαζόμαστε για τις εκλογέ του χρόνου και με τον ε, προεπιλογισμό μας σχεδόν δεν λάβαμε ε, τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για πρώτη φορά βέβαια λάβαμε τον έλεγχο ε, της διπραγμάτευσης. Σκεφτόμουν λοιπόν, εάν είχε περάσει αυτός ο κανόνας το 50 1, τι θα γινόταν με τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Θα ήθελα λοιπόν οι χώρες που έχουν αυτόν τον κανόνα του 50 να μας βοηθήσουν. αλλά και από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες. Οι περισσότερες έχουν ένα εκλογικό σύστημα του όποιος περάσει πρώτος ένα συγκεκριμένο ε, ε, ποσοστό κερδίζει. Και αυτό τελικά έχει θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now Joachim from the IT Electoral Commission. Από την εκλογική ε, ομάδα της ΑΙΤΙΣ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, οργανωτές και τις οργανώτες της διάσκεψης αυτής που έχουν εδώ ε, φέρει έγκριτες προσωπικότητες ε, που παρατηρούν εκλογές, οργανώνουν εκλογές. καθώς επίσης και ερετούς. δεν θέλω να μιλήσω για πολλή ώρα, αν και ε, πραγματικά εγώ είχα προετοιμάσει ένα λογίδριο για να, σας, ε, να μοιραστώ μαζί σας ε, τις εμπειρίες που έχουμε στην ΑΕΤ κυρίως βάσει των εκλογών του 2017 και του 2000, συγγνώμη, 2016 και 2017. Έχω εδώ βέβαια ένα έγγραφο μαζί μου, το οποίο σας έχω αφήσει και στην είσοδο ε, και το οποίο σας καλώ να διαβάσετε έτσι ώστε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Και περνώ άμεσα σε μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να διατυπώσω προς το πάνελ. Ιδίως ε, δε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρατήρηση Υπάρχουν καινοτομίε που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό που σας έδειξα, που έχουν καταγραφεί και στο νομοσχέδιο που έχουμε προετοιμάσει. Πρόκειται λοιπόν για μια μετεκλογική διαδικασία και οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν ε, την αντίδραση στις συστάσεις ε, της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης στη χώρα μου. Τώρα έχει υποβληθεί στην εκτελεστική ε, εξουσία ε, αυτό το, αυτή η πρόταση έτσι ώστε να περάσει στο Κοινοβούλιο. Και ερωτώ πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλίσει ότι σε αποδεκτό χρονικό όριο θα, γίνουν, ε, θα ενσωματωθούν ε, αυτά τα στοιχεία στο νέο εκλογικό νόμο έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και να ισχύσουν στην εκλογική διαδικασία του 2019. Hello, Χάνα Ρόμπερτς, ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να τονίσω τη σημασία των ε, παρατηρητών που θα πρέπει να μιλούν ειλικρινώς ακόμα και σε περιπτώσεις συγκρούσεων. Αν δεν πούμε την αλήθεια, μπορεί να ενισχύσουμε αυτούς που χρησιμοποιούν τη βία και τον εκφοβισμό. Κινδυνεύουμε να τους δώσουμε περισσότερη εξουσία για να εδραιώσουν τη θέση τους. Αν δεν μιλήσουμε με το γλώσσα της αλήθειας, μπορεί όντως να δώσουμε την εντύπωση στην, στους πολίτες να, την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να εμπιστεύονται πια τους ελέγχους και τις δημοκρατικές δομές. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον λόγο μας για την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τομεί που μπορούμε να ενισχύσουμε τι πρακτικέ τη παρατήρηση εκλογών. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τι ε, τις ε, συζητήσεις πριν τις ε, εκλογές για να δούμε τι πάει καλά, που υπάρχουν προβλήματα, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να μας εμπιστευθούν ότι όντως είμαστε ειλικρινεί και μιλούμε με το, η γλώσσα της αλήθειας. Επίσης, η διαδικασία για τα, για τα αποτελέσματα. Πολλές φορές αυτό είναι το πιο προβληματικό σε μια εκλογή. Και αυτό που σημαίνει, συμβαίνει είναι ότι έχουμε κάποιες ε, αρχικές δηλώσεις μετά τις εκλογές και η πολιτική ηγεσία φεύγει και μετά αρχίζουν να, αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα με τα αποτελέσματα. Αυτές οι αρχικές ε, ε, δηλώσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και μπορεί να φανεί ότι φτάσαμε με παρατηρητές ε, από όλη τη χώρα, μιλούμε για όλα τα, όλες τις πτυχές των εκλογών, αλλά φαίνεται σαν να μην έχουμε τίποτα να πούμε στο πιο σημαντικό σημείο της όλης διαδικασίας, τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας. Οπότε θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να, να δείχνουμε ότι όντως μιλούμε, την αλήθεια σε, μιλούμε με την γλώσσα της αλήθειας σε πραγματικό χρόνο. Ευχαριστώ. Άντε από το Κροατικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων που οργανώσατε σήμερα αυτή την ε, διάσκεψη. Από χτε ε, ακούσαμε ήδη πολύ σημαντικά πράγματα και πραγματικά όλα αυτά μας βοηθούν πολύ για τη δημοκρατία, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Η κυρία Ματίας ε, ρώτησε ποια είναι τα, τι μπορούν να κάνουν ε, τα μέτρα που παίρνουμε κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών και θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές έγιναν στην Βοσνία Ριζεγοβίνη στις 7 Οκτωβρίου και κατεδείχθη η έλλειψη εξουσίας αυτών των αποστολών. Οι αποστολές που έρχονται στη χώρα θα πρέπει να γνωρίζουν τον εκλογικό νόμο της χώρας για να μπορούν να υποβάλουν εκθέσεις για την εκλογική διαδικασία και να δίνουν πραγματικά στοιχεία. Η Βοσνία ριζεγοβινη είναι μια χώρα που αποτελείται από τρεις ε, εθνότητες ε, και δύο βασικές οντότητες. Κατά τη διάρκεια της, ε, της εκλογής οι πολίτες εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Έχουμε και βοσνιακή μειονότητα. Είναι η τρίτη φορά που οι Κροάτες χάνουν τις εκλογές από την βοσνιακή μειονότητα. Και ο Κροάτης εκπρόσωπος εκλέγεται από Βόσνιους. Θα πρέπει λοιπόν στις εκθέσεις μας να λέμε τι ακριβώς έχει γίνει. Οι ε, αποστολές παρατήρησης θα πρέπει να λαμβάνουν και αυτά τα στοιχεία υπόψη τους, γιατί αυτό πραγματικά εδρεώνει την, ασ, την ανασφάλεια και την αστάθεια και, η Βοσνία, και μια ασταθής Βοσνία Ζεγοβίνη σημαίνει αστάθεια στην Ευρώπη. Ξέρω ότι ο κύριο Κάρτερ τα γνωρίζει όλα αυτά και βεβαίω δεν θα πρέπει να καταπατώνται οι συμφωνίε και οι εκλογικέ αποστολέ θα πρέπει να λαμβάνουν και αυτά τα στοιχεία υπόψη. Ε, σα ευχαριστώ πολύ. Η Λάουρα Καστέλτσα από την Ισπανία και από το Σενάτο. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σα χαιρετώ. Θα ήθελα και εγώ βεβαίως να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, ε, οργάνωσαν αυτήν την διάσκεψη που είναι τόσο, τόσο ενδιαφέρουσα. Έγινε λόγος ε, για τα στοιχεία τα οποία μπορούν να κλιμακώσουν τη βία στις εκλογές ε, και την, ε, ποια, μπορεί να είναι η θρελίδα ας πούμε, αυτών των ε, βιωτήτων, ταυτοποίηση προβλάτων που μπορεί να δημιουργήσουν σειράξεις και τα λοιπά. Εγώ πολύ συγκεκριμένη ερώτηση θέλω να θέσω. ποια πρέπει να είναι τα βήματα που είναι απαραίτητα για να λυθεί μια κατάσταση την οποία είδα εγώ ως παρατηρήτρια εκλογών ο πρόεδρο μια κυβέρνηση. διαλύει ε, μια βουλή ε, υποκυβερνητικού επίπεδου. Ε, ε, ε, πάβει όλους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης χωρίς να έχει όμως τις θεσμικές συνταγματικές διαδικασίες και αρμοδιότητες γι' αυτό. Ορισμένα μέλη αυτής της κυβέρνησης μπαίνουν στην φυλακή, βρίσκονται ακόμα σε προσωρινή κράτηση χωρίς να προβλέπεται συγκεκριμένη ημέρα, ημερομηνία δίκης. Αυτή οι επικεφαλείς συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων βρίσκονται βρίσκονται στην φυλακή, μερικοί βρίσκονται στην εξορία και δεν μπορούν παρά να κάνουν προεκλογική εκστρατεία από απολύτως μειονεκτική θέση. Ε, προεκλογική διαδικασία η οποία έφτασε ακόμα και σε ε, μια παράνοια και απόλυτο παροξισμό που ήταν η ε, απαγόρευση της χρήσης του κίτρινου ε, χρώματος γιατί παρέπεμπε σε μια συγκεκριμένη ιδέα. Εδώ εγώ ε, σας ε, περιγράφω την κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια χώρα της Ευρώπης. Αυτά συνέβησαν πριν από μερικούς μήνες. Επομένως, αν μιλάμε για πολιτική δημοπλωματία, θα πρέπει να μιλάμε ε, και για αντιδραστική δημοκρατία με την έννοια της αντίδρασης σε κάποια πράξη. Και τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ε, κυρία Καστέλς, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι παρακολουθήσαμε ε, μαζί ε, τα ίδια γεγονότα τα οποία εσείς περιγράψατε, αλλά η δικιά μου περιγραφή και η δικιά μου ανάγνωση θα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Ε, οι, οι στιγμές τις οποίες εσείς μεταφέρατε εδώ, από τη δικιά μου πλευρά και τη δικιά μου αφήγηση, θα ήταν τελείως διαφορετικές. Δύο ακόμα αγορητές θα πάρουμε. Σαμσουνιτόδο από, την, ε, ε, από μια μη κυβερνητική οργάνωση που ονομάζεται ε, Αφρικανική Νεολαία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατάγομαι από την Ιγυρία, μία από τις χώρες στην Αφρική, όπου θα γίνουν εκλογές μέσα στις επόμενες 127 ημέρες. Να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα. Αρχικά να ευχαριστήσω τον πρέσβη κύριο Τσάμπας για το σχόλιο του για την Ιγυρία, για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν τις εκλογές ε, στην Ιγυρία. Πρώτον, η τεχνολογία και η αγκαιρεότητά της. Δεύτερον, η συμμετοχή στην ε, ψηφοφορία που βλέπουμε στην Ιγυρία, όπου ουσιαστικά εξαγοράζονται ψήφοι από τους πολιτικούς. Ε, τρίτον, ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας. Κύριε Τσάμπας, στη δική σας ε, εμπειρία με τα θεσμικά όργανα στην Ιγυρία, είναι σημαντικό να δείτε τις ε, ε, υπηρεσίες ασφαλείας, το η τάση και το πιο σημαντικό εργαλείο για τις εκλογές και την καταστολή των εκλογών στην Ιγυρία είναι ακριβώς αυτά τα μέσα. Πρόσφατα είχαμε μια εκλογική διαδικασία που η αστυνομία απέτρεψε ε, τους ε, ψηφο, ορισμένους ψηφοφόρους που υποστήριζαν συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες να φτάσουν ε, στα εκλογικά κέντρα. Και εφόσον μιλούμε για την ασφάλεια και την ειρήνη, είναι πολύ σημαντικό ε, να λογοδοτούν και να είναι υπεύθυνε οι υπηρεσίε ασφαλεία. Και τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία και από πλευράς πολιτικών. Γιατί οι πολιτικοί ε, που προσπαθούν να παρακινήσουν τους νέους ε, προς βίες, ε, βία ξεσπάσματα, ποτέ δεν λογοδοτούν τελικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει λογοδοσία αυτών των πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τελευταία παρέμβαση. Η Ρωμάνα Χέτια ε, Κίτε από τη Σρι Λάνκα. Σίγουρα έχω ε, ε, διαβάσει λάθο το όνομά σα. Ελπίζω να καταλάβατε όμως περί ποιου πρόκειται. Ρωμάνα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα όσα είπατε και να σας μεταφέρω μια εμπειρία από την Ασία. Αυτή η βία μπορεί να διαχωριστεί σε δύο επίπεδα. Φυσικά, σε ένα επίπεδο η βία δημιουργείται από κάποιους πολιτικούς και η υπόλοιπη βία ξεκινάει από μόνη της από τους ψηφοφόρους. Φυσικά υπάρχει εδώ ο ρόλος ε, της διεθνούς κοινότητας για να αποτρέψουμε σε ένα βαθμό τη βία με την οικοδόμηση ενός ε, σωστού συστήματος και οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς το εκλογικό σύστημα, τότε αυτή την ε, φυσική βία μπορούμε να την αποτρέψουμε σίγουρα. Υπάρχει αυτή η εμπειρία, ειδικά στη χώρα μου. Και υπάρχει και σύστημα ε, καταγραφής των ψηφοφόρων μέχρι και επίλυσης διαφορών. Με αυτά τα μέσα σίγουρα μπορεί να μετριαστεί και να αποτραπεί η φυσική βία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι περιφερειακοί φορείς μπορούν ε, να στηρίξουν ε, τους φορείς που αναλαμβάνουν αυτή την αρμοδιότητα. Βέβαια, μετά είναι και το σκέλος των πολιτικών που υποκινούν τη βία. Υποκινούν τη βία λοιπόν επειδή υπάρχει ένα σαθρό σύστημα. Εάν το διορθώσουμε, σίγουρα μπορούμε να αποτρέψουμε σε ένα βαθμό αυτή τη βία κατά τη δική μου εμπειρία. Ευχαριστούμε. Τώρα θα πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να μιλήσουν όλοι οι πανελίστες ε, Ελπίζω οι διερμηνείς να μας δώσουν, λέει η Πρόεδρος, λίγο χρόνο. Και νομίζω ότι πρέπει να πείτε εσείς αυτή τη στιγμή ποια είναι η σύσταση, η καλύτερη που μπορείτε να κάνετε ε, αυτή τη στιγμή. Οι κυρίες πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω ε, στην κυρία προηγουμένω στην βουλευτή η οποία μίλησε για τις γυναίκες μεσολαβήτριες που κάνουν δηλαδή αυτήν την ε, ε, μεσολάβηση είναι, εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο πρόβλημα ε, στην Αφρική. Όταν ε, ε, βλέπουμε αντιπροσωπείες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν διαμεσολάβηση ειρήνευση, οι γυναίκες είναι απούσες. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το θυμάται αυτό και να δράσει με τρόπο ώστε να υπάρξουν γυναίκες μεσολαβήτριες. Επίσης, μετά τις εκλογές, ε, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εκπροσώπων της να μείνει και μερικές μέρες μετά τις εκλογές τουλάχιστον δύο μέρες μετά τις εκλογές ε, ε, να βοηθήσετε τη σταθεροποίηση της χώρας πριν σηκωθείτε, τα μαζέψετε και φύγετε, λέει ο Μιλήτρια γιατί οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα ακούσουν τον τοπικό πληθυσμό, αλλά θα ακούσουν όμως την διεθνή ε, κοινότητα. Το έχουμε δει αυτό, είναι σημαντικό να παραμείνετε δηλαδή επί τόπου, τουλάχιστον δύο μέρες. Και κάτι τελευταίο ένας ε, ε, ε, επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης στην Κάνα είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ στη ζωή μας αναλάβει δέσμευση τέτοιου είδους. Πρέπει στις εκλογές να νοιαστείτε και για τους ανθρώπους που πραγματικά είναι σημαντικοί να ξεκινήσετε από χαμηλά, να ξεκινήσετε από τη νεολαία, από τις, από τις γυναίκες Πρώτη φορά, πρώτη φορά είδαμε ε, κάποιους ε, που πραγματικά να μιλάνε μαζί μας ε, και να μεταφέρουν το δικό μας μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπλακεί η νεολαία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τσάμπας. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε και μία συγκεκριμένη ερώτηση προς εμένα από τον νεαρό φίλο μας από την Ενιγυρία, καθώς επίσης και από την κυρία από το Μαλάουι, την εκλογική επιτροπή του Μαλάουι. Ναι, βεβαίως πρέπει να εστιάσουμε στα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Μόλις γύρισα από την Αμπούτζα και ακριβώς κάναμε μία επίσκεψη στην ε, Νιγηρία. η Νιγερία μεταξύ των δύο ε, εκλογών ε, και ήρθαμε σε επαφή με τους επικεφαλείς των security agencies. Είδαμε τι έγινε το 2015. Είχαμε, όλοι δέχτηκαν, παραδέχτηκαν ότι ήταν ασφαλής η διαδικασία. Δεν ήταν εκφοβιστική η παρουσία των ε, αρχών ασφαλείας. Ε, χρειαζόμαστε την ε, παρουσία των ανδρών ασφαλείας και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και μια διακριτική παρουσία του στρατού. αυτό αυτό θέλουμε να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες ασφαλείας να κάνουν. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες της Νιγηρίας, ε, κυρίως εκεί που τα προβλήματα της ασφάλειας είναι μεγαλύτερα, ε, το διακύβευμα είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αρκετά ασφαλές έτσι ώστε ας πούμε στον, ε, στα βορειοανατολικά να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν οι άνθρωποι με ασφάλεια ας πούμε εκεί που δράει Μποκοχαρά Πρέπει με κάποιο τρόπο να ε, διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής. Ε, όσον αφορά τη λογοδοσία, γνωρίζετε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ε, να ε, υπάρξει μια εξειδικευμένη επιτροπή η οποία ε, θα έχει την δυνατότητα διερεύνησης αλλά ακόμα και προσαγωγή στα δικαστήρια περιπτώσεων παραβίαση του εκλογικού νόμου. Αυτό είναι καλό γιατί η κοινωνία θα το δεχτεί αυτό και θα το δεχτεί με ανακούφιση. και βεβαίως θα πρέπει ε, να υπάρξει ε, συνένεση εντός του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να προωθηθεί ε, αυτή η νομοθεσία. Και αυτό θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 50 1 ή ο, αυτός που έχει μία ψήφο παραπάνω κερδίζει. Θα συνεχίσουμε να το συζητάμε. Στην Δυτική Αφρική το 50 1 έχει γίνει δεκτό σαν περιφερειακός κανόνας λόγω ε, κάποιων ιδιαζουσών καταστάσεων που επικρατούν στην περιοχή. Ε, δυσχέρεια επιτεύξης ε, εθνικής συνένεσης. και όντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου ε, βλέπουμε χειραγώγηση έτσι ώστε ε, να παραμείνει κάποιος στη θέση του έστω και αν δεν έχει φτάσει στο 50% και έστω και αν είναι δηλαδή μειοψηφία. Σε πολλές ε, χώρες υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα πρότεινα λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει coupling των εκλογών Ε, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ε, ακόμα και σε επίπεδο όχι μόνο των βουλευτικών εκλογών, αλλά και των προεδρικών. Οι χώρες λοιπόν οι οποίες δεν έχουν το σύστημα θα πρέπει να το δούνε. Γιατί είναι πάρα πολύ ε, προβληματικό να έχουμε εκλογές συνέχεια κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσάμπας, επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Θα μιλήσω γενικώ και λίγο έντονα, γιατί πρέπει να πω ότι κάποιος θεωρεί ότι ο παρατηρητής εκλογών είναι διαιτητής εκλογών. Θέλει να δώσει φάουλ και προσπαθεί να θέλουν να ρυθμίσει τον αγώνα, αλλά αυτό δεν είναι ο ρόλος. Δεν είναι δική μας η δημοκρατία. Η δημοκρατία ανήκει στους πολίτες της χώρας. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και ο πραγματικός ρόλος είναι να κρατήσουμε έναν καθρέφτη ο οποίο αντικατοπτρίζει τι γίνεται ακριβώ. Και οι εκλογέ είναι η χρονική στιγμή που μπορεί κανεί να αξιολογήσει τι είναι η δημοκρατία, πόσο διαφανής είναι, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, ποιο συμπεριλαμβάνεται και ποιο όχι. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, όπω υπόθηκε, είναι ότι όντω πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα τη αλήθεια, γιατί αλλιώ δεν είσαι αξιόπιστο και καλό καλή τυπίστη παίχτη του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν και οι εθνικοί οργανισμοί που υπάρχουν, οι εθνικοί παρατηρητέ, οι απόψει των ανθρώπων που ζουν εκεί και γενικώ το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται μια κατάσταση. Όταν ε, σεβόμαστε όλα τα επίπεδα, όπω ε, υπόθηκε, τους ε, μηχανόβιου ή τους διάφορους άλλους οργανισμούς που υπάρχουν και που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, μπορούμε να δείξουμε πραγματικά τι γίνεται μέσα σε μια δημοκρατία και μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να πιστέψουν στο μέλλον αυτής της ε, δημοκρατίας. Αυτό κρατάει τους πολίτες εντός του πολιτικού συστήματος και δεν ε, κλείνουν προς την βία. Πρέπει λοιπόν να τα εγγράψουμε όλα αυτά στην όλη διαδικασία για να έχουμε τελικά καλό αποτέλεσμα. Ο κύριος Χάβιστο. Ευχαριστώ. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε κάποιε. Καταρχάς, αυτό που είπε η κυρία Πόστ, η ανασφάλεια που υπάρχει μετά τις, ε, ε, ε, πριν τι εκλογέ. και για το πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει. Αν δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική διαδικασία, α πούμε, και δεν υπάρχει ηρεμία πριν τι εκλογέ, τότε προφανώς κάτι πήγε στραβά. Βεβαίως, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να παραμείνουν στην όλη διαδικασία και αν προκύψουν προβλήματα είναι σημαντικό να υπάρχουν. Τώρα για τους ενδιάμεσους, για τις γυναίκες ε, διαμεσολαβήτριας, ε, έχουμε και στην ε, Ευρώπη το σκανδιναβικό δίκτυο που γυναικών διαμεσολαβητών. Τώρα για την εξαγορά ψήφων ο συνάδελφος από την Ιγυρία το είπε αλλά εγώ πρόσφατα ταξίδεψα στα Δυτικά Βαλκάνια και πολλοί νέοι μου είπαν ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα που μία ψήφος σου δίνει δουλειά. Το κράτος, ε, ε, το πολιτικό κόμμα που ε, έχει την εξουσία ουσιαστικά ελέγχει και τις θέσεις εργασίας. Πραγματικά εμένα με εξέπληξε αυτό. Δυστυχώς αυτές οι πρακτικές εξακολουθούν. Και μετά από τον, για τον κύριο από τη Σρι Λάνκα Πρόσφατα κάνατε ένα πολύ καλό σεμινάριο στο Κολόμπο και μιλούσε για την διαφάνεια και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αν η αξιολόγηση είναι αυτό που πρέπει να γίνει, ας, γίνει αυτό. Ήταν πραγματικά ένα πολύ επιτυχές σεμινάριο, γιατί όντως η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Δύο ώρες είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε, δεν αποφασίζουμε εμείς ε, για τη χρονική διάρκεια της συνεδρίας. Ε, έτσι είναι και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ε, ξεκινώντας από την συζήτηση που είχαμε λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε ε, να εξάγουμε συμπεράσματα που μπορούν να αποβούν ε, χρήσιμα σε όλους. Θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο εκ των προτέρων εξάντε για περισσότερο διάστημα, σε περισσότερο βάθος ε, να έχουμε περισσότερες επαφές με το σύνολο των ε, φορέων και πρωταγωνιστών σε, της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Εξάντε λοιπόν ε, συνεργασία και μεταξύ των διαφόρων φορέων της διεθνούς κοινότητος και με αυτούς που ασχολούνται με την ασφάλεια και την ειρήνη ενδυνάμωση της διασύνδεσης ανάμεσα στην παρατήρηση και την αρρωγή στη διάρκεια των, ε, και στα πλαίσια των εκλογών και κινητοποίηση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν που ενδεχομένως είναι και λίγο διάσπαρτοι και ελαφρώς ασυντόνιστη. Καλύτερο συντονισμός ας πούμε ανάμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ηνωμένων Εθνών και την ε, Αφρικανική Ένωση ε, συνέργειες και συντονισμός ο οποίος έχει υπάρξει μεταξύ των τριών ε, θεσμικών φορέων που μπορούν να, μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα και για ε, περαιτέρω συντονισμό και συνεργασία. Προκύπτει από τα όσα ε, υπόθηκαν η ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση ε, σε μέσο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Δηλαδή όχι να παραμείνουμε μόνο στη διάρκεια των, ε, της προεκλογικής ή μέχρι τη μέρα των εκλογών, ε, αλλά και μετά την καταμέτρηση. γιατί και αυτό αποτελεί μέρος της εργασίας μας και του ελέγχου των δημοκρατικών συστημάτων η πρόληψη ε, της ε, βίας ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να βασίζεται σε μέτρα τα οποία θα έχουν ληφθεί πριν από την παρατήρηση των εκλογών. Ωστόσο, οι παρατηρητές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα, θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν και καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν επιτόπου και στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και βεβαίως οι πολιτικοί υπεύθυνοι των ε, ομάδων παρατήρησης ίσως θα πρέπει να έχουν και μεγαλύτερη κατάρτιση όσον αφορά ε, τις συγκρούσεις. Γιατί είδαμε ότι αυτό το σκέλος ε, δεν είναι πολύ αναπτυγμένο. Αυτό που είναι σαφές νομίζω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιολογήσει με σωστό τρόπο τις ε, χώρες και τις ε, συγκεκριμένες ε, χρονικές στιγμές που θα στείλει τις ε, αποστολές σας. Ε, ε, οι πόροι μας δεν είναι ατελείωτοι, άρα οι αποστολές δεν μπορεί να είναι ατελείωτες. Αυτό είναι σαφές και επομένως θα πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή της χώρας στην οποία θα γίνει η παρατήρηση, γιατί μερικές φορές δεν αξίζει τον κόπο να πάμε σε μια χώρα, ενώ υπάρχει άλλη χώρα η οποία πράγματι έχει δείξει συγκεκριμένα δείγματα γραφής βούλησης για ποιοτική εκλογική ε, αναμέτρηση. Ε, Βεβαίω κατανοώ ότι όλοι έχουμε και κάποιες δημοκρατικές δεσμεύσεις, διορθώνω κάποιες διπλωματικές ε, δεσμεύσεις κλπ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, γιατί υπάρχουν σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, που δεν χρειάζεται καν διερευνητική αποστολή. Δεν κάνουμε δημοσιογραφία εδώ, πρέπει να προετοιμάζουμε την εκλογική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας αποχαιρετήσω όλους και να σας πω ότι αν θέλετε να συμμετάσχετε στο επόμενο πάνελ Ε, αν θέλετε μάλλον να ε, ε, πάτε στην, στο άλλο πάνελ για τη συνεργασία Αφρικανικής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάτε στον τέταρτο όροφο όπου 11 και 20 θα ξεκινήσει μια άλλη διάσκεψη, ένα άλλο πάνελ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο πάνελ όμως θα λάβει χώρα εδώ. Δηλαδή μπορείτε να μείνετε και σε αυτή την αίθουσα.